La séance est reprise. Συνεχίζουμε τη συνεδρίαση. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας εκεί που τις αφήσαμε χτες. Να σας πω ότι θα εξετάσουμε τις κατηγορίες ως εξης ένα 1α, μετά τα ειδικά μέσα, μεταφορά προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όπως συμφωνήσαμε χτες. τέσσερα πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις. Άλλες, άλλα, άλλα τμήματα και πληρωμές. Για την 1α η Γενική Συγγήτρια έχει μία διευκρίνηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως σας είπα έχω μια, ένα μικρό σχόλιο. Μια τεχνική αλλαγή μετά από τόσες αλλαγές ε, και διαπραγματεύσεις άλλαξαν πολλές φορές τα νούμερα. Στον τελευταίο πίνακα ξεχάσαμε λοιπόν μια γραμμή να αλλάξουμε. Στο πρόγραμμα 090303 στο τμήμα για τις υποχρεώσεις που ξεπερνούν την πρόταση, που υπερβαίνουν το ποσό της πρότασης της επιτήρησης above DB, αντί για 6 να βάλουμε 10 εκατομμύρια στο παράτημα που έχετε μαζί με τη συμφωνία για την κατηγορία 1α. Επαναλαμβάνω 090303 είναι το Promoting Interoperability Sustainable Deployment Operation Upgrading of Terms European Digital Service Infrastructure and uh, coordination at European level. Αντί για 6 βάζουμε 10 εκατομμύρια και μετά ψηφίζουμε. Donc une, une correction. Διόρθωση είναι. Γενναιόδορη διόρθωση. Ο κύριος Ντιπρέ έχει το λόγο. Πρόεδρε. Χτες είχα πει ότι στην χτεσινή ψηφοφορία δεν είχαμε προβλήματα. Ενδεχομένως να είχαμε σήμερα, ωστόσο, για το 1α και για την κατηγορία 4. Δεδομένων των προσπαθειών της εισηγήτριας και θέλω να την ευχαριστήσω δημοσία για τις προσπάθειές της, αλλά και από τις προσπάθειες του συντονιστή ΕΛΚΑ, κάποια από τα θέματα που μας δημιουργούσαν προβλήματα επιλύθηκαν. Άρα μπορώ να σας αναγγείλω ότι και για το 1α και για το 4 οι αντιρρήσεις που είχαμε έχουν αρθεί και ευχαριστώ όλους όσοι επέτρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο. Είδατε τώρα που ξεκινάει η μέρα κύριε Ντεπρέ. Προχωρούμε. Κατηγορία 1α. Πρώτη υπομάδα, αποκατάσταση του σχεδίου προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις όπως είχαν προταθεί δηλαδή από την Επιτροπή στην αρχική, στο αρχικό στάδιο. Οι λεπτομέρειες είναι στο παράτημα πίνακα 1. Ψηφίζουμε υπέρ της έγκρισης τροπολογίας. Ευχαριστώ. Κατά. Τέσσερις. Κατά. Η ομάδα των τροπολογιών εγκρίνεται. Δεύτερη υποομάδα διατάξεις που επαναφέρουν, που φέρουν πιστώσεις υπεράνω των προβλεπωμένων από την Επιτροπή. Παράδειγμα πίνακας 2. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τέσσερις κατά. Εγκρίνεται και η ομάδα αυτή τροπολογιών. Προχωρούμε στις υπόλοιπε ψηφοφορίε, τροπολογίε που δεν έχουν καλυφθεί από τι συμβαστικέ προτάσει. 010201. Πρώτη τροπολογία. 796. Η συγγήτρια είναι κατά. Ψηφίζουμε υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται η τροπολογία. Στην ίδια γραμμή. 527 τροπολογία. Η εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Όχι. 619 6-19 τροπολογία. Η εισηγήτρια είναι κατά υπέρ της τροπολογίας. Je vous remercie. Baissez les mains. Avis contraire. Κατά. Baissez les mains. Abstention. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται. 02-02-01 γραμμή. 42-11 τροπολογία. Η είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται. Γραμμή 020202. Τροπολογία 755. Και 4212. Η εισηγήτρια είναι κατά ποιήν υπέρ. Κάτω. Τα χέρια. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία. Γραμμή 0403-0101, τροπολογία 1018. Ε, ο εισηγητής είναι κατά. Η εισηγητή, συγγνώμη, κατά ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται. Στην ίδια γραμμή, 759 τροπολογία και 4216. Με το ίδιο αντικείμενο. Η εισηγήτη είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται. Στη γραμμη 02, 0802-03-01 815 τροπολογία και 4273 ίδιες. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται η τροπολογία. Γραμμή 08020302, τροπολογία 816 και 4274, η 3 είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται. απορρίπτεται, Τροπολογία 859 και 4317. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές καμία απορρίπτεται γραμμή 0803-0102 το απολογία 670 η εισηγήτρια είναι κατά ποιοι είναι υπέρ ευχαριστώ κατά αποχές καμία απορρίπτεται η τροπολογια 5524 55-24 η τοπολογία η εισηγήτρια είναι κατά ποιοι είναι υπέρ κατά εποχές καμία απορρίπτεται το γραμμή 08040101 τροπολογίες 666 και 874 η εισηγήτρια είναι κατά ποιοι είναι υπέρ κατά εποχές δεν υπάρχουν απορρίπτεται 08-04-01-02 668 εισηγητής είναι, εισηγητή είναι κατά ποιοι είναι υπέρ ευχαριστώ κατά απαχές καμία 2 απορρίπτεται 09040302 04 το 02 821 και 4279. Η είναι κατά ποιοι είναι υπέρ Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται η τροπολογία. Γραμμή 12.03.01. Τροπολογία 3.57. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Όχι. Απορρίπτεται. Στην ίδια γραμμή έχουμε την τροπολογία 1005. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ? Ευχαριστώ κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται και ότι εγκρίνεται διορθώνει ο μιλητής, αλλά ας κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. πέρα στις εγκρίνεται 17 υπέρ 14 κατά 02 01 8 51 και 43-09 η εισηγήτρια είναι κατά ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Γραμμή 15.02.01.02. Δύο τροπολογίες, 853 και 43.11. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Τρεις. Απορρίπτεται η τροπολογία. Στην ίδια γραμμή τροπολογίες 825 και 4283 με το ίδιο αντικείμενο εισηγείται είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας, των τροπολογιών αυτών. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δύο. Η τροπολογία απορρίπτεται. Στη γραμμή 15.03.02 τροπολογίες 8.22.42.80. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. αποχές καμία απορρίπτεται. Στη γραμμή 02010601 η τροπολογία 4039. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία. Δύο. Απορρίπτεται. Γραμμή 020201. Δύο τροπολογίε. Η 4211 και η 754. Η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. αποχέ. Καμία. Απορρίπτεται η τροπολογία. Η ίδια γραμμή, η τροπολογία 926. Αντικείμενο θετικής Αποψη της ηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην ίδια γραμμή τροπολογία 386. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία. Στην 020202 γραμμή, η πρώτη τροπολογία, δύο τροπολογίες, 755 και 4212, η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην ίδια γραμμή 360 τροπολογία. Η εισηγήτρια εδώ είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Τρει αποχέ. trois abstentions. L'amendement est... Τρεις αποχές. Εγκρίνει η τροπολογία. Γραμμή 0204-0203. Τροπολογία 659. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία εδώ. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Στο ΕΛΚ φαίνεται ότι υπάρχει ένας που είναι παραπάνω από αυτούς που δικαιούνται να ψηφίσουν. Εντάξει. Καλή η πολύ, αλλά μέχρι σωρίου. Απορρίπτεται η τροπολογία. 16 υπέρ, 18 κατά. 04, 03, 01, 04. Πρώτη τροπολογία. 650. Ε, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Οποχές. Εγκρίνεται. Στην ίδια γραμμή. 4.134. Ε, κατά είναι η συγκήτρια. Ποιοι ειναι πέρα υπέρ. Κατά. Αποχές. 03 04-03-01-03. Τροπολογία 361. Η συγκήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Ή ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται η τροπολογία. 17 υπέρ, 14 κατά. 04, 03-01-04. Πρώτη τροπολογία 40-43. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας. Ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές δεν έχουμε. Απορρίπτεται. 387. Υπέρ εισηγήτρια. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τρεις. Αποχές. Δύο. Εγκρίνεται. Ίδια γραμμή. 4.074 κατά εισηγήτρια υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω. Απορρίπτεται. 0403-0105. Τροπολογία 4041. Κατά εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν έχουμε. Απορρίπτεται 0403-0201, τροπολογία 388, υπέρ εισηγήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται η τροπολογία 17-17 είναι το αποτέλεσμα. 17-17 απορρίπτεται. Τροπολογία 40-73. Κατά εισηγήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 04-03-02-02, τροπολογία 364. Υπέρ παρακαλώ, υπέρ η Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ, 14 κατά. 04, 03, 02, 03. Τροπολογία 41, Κατά η συγκήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές δεν έχουμε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 365. Υπέρ συγγήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γραμμή 06 06-02-01-01, 01 τροπολογία 472 και 654 που έχουν το ίδιο αντικείμενο, κατά εισηγήτρια, υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 08 Απορρίπτεται. 08-02-02-01, τροπολογία 40 40-54, κατά εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 08-02-02-03, 661. Κατά εισηγήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην ίδια γραμμή, τροπολογία 385, υπέρ εισηγήτρια. Υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, 2. Εγκρίνεται. Γραμμή 080203. Τροπολογία 368. Υπέρ η συγκίτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 08020301. Τροπολογία 392 340. Κατά η συγκίτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. δύο Απορρίπτονται. Τώρα 392 υπέρ. Πριν ήταν 815 και 4340. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις εγκρινεται Εγκρίνεται. 16-15 και δύο εποχές. 43-40 υπέρ η εισηγήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές καμία. Α, δύο. Εγκρίνεται. 08, 02, 03, 02, τροπολογία 816 και 4274. Κατά η εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 2. Απορρίπτεται. Γραμμή 08-02-03-03. Τροπολογία 110. Και υπάρχει εδώ και προφορική τροπολογία της εισηγητρίας. Με την επιφύλαξη αυτής της προφορικής λοιπόν είναι υπέρ εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές δεν υπάρχουν. Εγκρίνεται λοιπόν με την προφορική τροποποίηση. 08, 02, 03, 06, 369. Υπέρ εισηγήτρια. Υπέρ. κατά αποχές όχι εγκρίνεται 43.99 υπέρ η υπέρ παρακαλώ κατά αποχές δεν έχουμε εγκρίνεται 080204 Τροπολογία 818 και 4276. Υπέρ η συγγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 21 ψήφοι κατά, 2 υπέρ. 08, 03, 01, 02, τροπολογία 670. Κατά η συγκίτρια. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δύο. Απορρίπτεται. Γραμμή 090302. Τροπολογία 4128. Κατά η συγκίτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Όχι. Απορρίπτεται. 09-03-03. 264 τροπολογία. Υπέρ η συγκήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γραμμή Γραμμή τροπολογία 40-55. Κατά η συγκήτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω. Απορρίπτεται. 10.03.01. Τροπολογία 669. Κατά εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 14.03.01. Τροπολογία 40.46. Κατά η εισηγήτρια. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. 14.04.01, τροπολογία 41.31, υπέρ, εισηγήτρια, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 15.02.01.01, πρώτη τροπολογία 851 και 4309. Υπέρ η εισηγήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 16 κατά, 15 υπέρ. Τροπολογία 43-38 στην ίδια γραμμή. Υπέρ η εισηγήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γραμμή 15.02.01.02. Τροπολογία 853 και 43.11. Είναι υπέρ η συγκεντρία είναι υπέρ παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 18 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. Γραμμή 150203, τροπολογία 266, υπέρ η συγκήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15.02.03.266 υπέρ. Επαναλαμβάνει την ίδια ψηφοφορία ο πρόεδρος. Α, συγγνώμη λέει. Συγγνώμη. Θα ήθελα να επαληθεύσουμε. 266 είναι υπέρ η συγκήτρια. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται, ναι. 24.02.01. Τροπολογία 41.29. Κατά η υπερ Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. 32040301. Τροπολογία 111. Με μια προφορική τροπολογία. Ίδια με την προηγούμενη που εγκρίναμε πριν από λίγο. υπέρ η συγκήτρια. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται. Τελειώσαμε λοιπόν με την κατηγορία 1α. Περνάμε τώρα στα ειδικά μέσα. για τα ειδικά μέσα. Έχουμε χωριστές Τροπολογία 79-83. Κατά η συγκίτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Θέλετε το λόγο κύριε Ντεπρέ. Παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Ντεπρέ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Ομολογώ ότι με εκπλήσει κάπως η μεγάλη αύξηση των μέσων που προβλέπονται σε αυτήν την γραμμή του προπολογισμού. Δεν έχω βέβαια μπροστά μου τα χαρτιά, αλλά από ό,τι θυμάμαι στο σχέδιο προπολογισμού της Επιτροπής ήταν 25 εκατομμύρια. Και εδώ περνάμε στα 150 εκατομμύρια. Με εκπλήσει η σημαντική αυτή αύξηση εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι υπερβολή σε σχέση με τον ρυθμό χρήσης των κονδυλίων τις προηγούμενες χρονιές. Προσοχή λοιπόν, γιατί είναι, υπάρχει μια τροπολογία της Επιτροπής Γυναικών που προβλέπει ένα χαμηλότερο ποσό. Ομολογώ ότι με εξέπληξε το μεγάλο αυτό ποσό δεδομένης της κατάστασης και θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρακαλώ. Η συγγήτρια. Α, η πρώτη κομισιόν. Α, όχι, όχι, ναι, τη δικιά σου την άποψη την ξέρω, γι' αυτό δεν ρωτάω, λέει στην εισηγήτρια ο κύριος Δεπρέ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο θα μιλήσει εκ μέρου της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι εκτιμήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτές που αναφέρονται στο σχέδιο προπολογισμού 2015 και που υπενθυμίσαμε και χτες. Πρόκειται για εκτιμήσεις προσεκτικές μεν, αλλά ρεαλιστικές. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μείνει στις εκτιμήσεις της. Ορίστε. Αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Ντεπρέ, άρα συμφωνεί μαζί σας, έτσι. Ναι, η Επιτροπή λέει ότι είναι σωστό, αλλά εμένα με εκπλήσει το ποσό που ζητάμε να αυξήσουμε, θα έπρεπε να είχαμε μια πιο προσεκτική και περιορισμένη αύξηση. Να ψηφίσουμε τον γυναικών την τροπολογία που μιλάει για 50 εκατομμύρια, διπλασιάζεται το ποσό, ενώ με τα 150 εκατομμύρια το πολλαπλασιάζουμε επί 6. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν ένα πολιτικό μήνυμα, αλλά μου φαίνεται υπερβολή. Πρόεδρος η παγκοσμιοποίηση σημαίνει αυτό ότι θα έχει τρομερές συνέπειες με έξι φορές παραπάνω το ποσό. Παρακαλώ κύριε Γιάλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι θέλουμε να επανέλθουμε στο αρχικό ποσό ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν αρκετά χρήματα στη διάθεσή τους και να μην πρέπει να περιμένουν 18 μήνες για να αποζημιωθούν. Αυτό ζητάμε μόνο. Δεν ζητάμε αύξηση ουσιαστικά, ζητάμε ανάκτηση του αρχικού ποσού. Πρόεδρος, υπενθυμίζω ότι εδώ είμαστε για να ψηφίσουμε, ότι η συζήτηση έχει λήξει. Συνεπώ. ψηφίστε τις τροπολογίες. Γραμμή 040401, τροπολογία 7983 λοιπόν, κατά η Γενική Συγήτρια, υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4258. Είναι ίδια, άρα δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Τώρα, τροπολογία 7401. Υπέρ. Η συγκεντρία υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα την τροπολογία 62-10. Α, όχι, καταπίπτει. Εφόσον εγκρίθηκε 74-01. Γραμμή 13-06-01 τώρα. Τροπολογία 84-79. Κατά η συγκήτρια. Υπέρ. Τρεις

και οι επόμενες καταπίπτουν. Σχόλια τώρα. Στα σχόλια 040401. Έχουμε την τροπολογία 6... Δηλαδή 11 λέει ο πρόεδρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελειώσαμε έτσι και με τα ειδικά μέσα. Περνάμε τώρα στις μεταφορές πιστώσεων. Από το 3 στο 10. Χτες αποφασίσαμε να αναβάλουμε τη ψηφοφορία. Τώρα όμως μπορούμε νομίζω. Θέλετε το λόγο, κύριε Χορμάγερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χρωστάω μια απάντηση στους συναδέλφους από χτες. Γιατί υπήρξαν και πολύ προσεκτικές ε, τοποθετήσεις. Πλέον έχουμε μια πλήρη συμφωνία και με βάση αυτή τα έξοδα, οι δαπάνες που αφορούν μετακομίσεις και ταξίδια, κτίρια και IT, πληροφορία, Ε τεχνολογία πληροφοριών, θα πάνε στο AD, ως όλα τα δα, όλες τις δαπάνες αφορούν το προσωπικό, βαρύνει την Κομισιόν. Το πρόβλημα είναι ότι αν κάποιος κάνει ένα ταξίδι πρέπει να αιτηθεί τα χρήματα αυτά στην Κομισιόν και είναι περίπλοκο αυτό το σύστημα. γιατί όλα αυτά αφορούν επιτόπου την, την, τα, τα κτίρια, τους ανθρώπους, ε, τη, την πληροφορική, οπότε όλα, για απλούστευση ε, ε θα μειώσουμε τις γραμμές από 15 σε 3. Ε, το Συμβούλιο δεν θέλει να γίνουν περικοπές. Αν προκύψει κάτι που θα είναι, αν το Συμβούλιο προσπαθήσει να μειώσει με κάποιον τρόπο τα κονδύλια, εγώ θα πρότεινα να κάνουμε μια ψηφοφορία εδώ στο Κοινοβούλιο, αν και κανονικά αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον είναι ότι υπάρχει συμφωνία, το Συμβούλιο δεν προτίθεται να κάνει περιορισμούς, να κάνει μειώσεις, Απλά πρόκειται για μια απλοποίηση, μια απλούσταση των διαδικασιών. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά όσον αφορά το ε, προσωπικό. Ωραία. Άρα, εντάξει, κατά εισηγήτρια. Παραμένουμε σε αυτό. Έτσι ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ, τη τροπολογία αυτή μεταφορά πιστώσεων. Κατά εισηγήτρια, είπαμε. Α, υπέρ, υπέρ εισηγήτρια τώρα. Υπέρ. Υπέρ εισηγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ, αυτή τη τροπολογία. Κατά. Κανείς, ούτε αποχές. Ωραία, τους απεφασίστε. Και περνάμε στην κατηγορία 4. Κατηγορία 4 λοιπόν. Έχουμε πρώτα απ' όλα ψηφοφορία επί ομάδων τροπολογιών που θέλουν να επανέλθουν οι πιστώσεις στο επίπεδο που τις είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο προπολογισμού της. Πρόκειται για τον πίνακα 7. Πρόκειται για ποσά κάτω από τα ποσά που είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υπέρ η Γενική Εισηγήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ναι. Αποχές. Δεν έχουμε. Εγκρίνεται η τροπολογία αυτή. Δεύτερη υπομάδα λοιπόν για να επανέλθουν οι πιστώσεις στο επίπεδο που είχε προτείνει η Επιτροπή Πρόκειται για τον πίνακα 8 του παραρτήματος. Είναι υπέρ η Γενική Συγκήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. 5 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία αυτή. Και τρίτη υπομάδα για να έχουμε πιστώσεις πάνω από το επίπεδο που είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πίνακας 9 στο παράρτημα δηλαδή. Η Γενική Συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ, παρακαλώ, της τροπολογίες αυτής. Κατά. Δεν έχουμε αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στις υπόλοιπε τροπολογίε που δεν καλύπτονται δηλαδή από τι συμβαστικέ. Υπάρχουν τέσσερι για τη γραμμή 01-03-02, 19-03-01-02, 19-03-01-03 και 19-03-01-04. Τις τέσσερις αυτέ τροπολογίε θα μπορούσαμε να τι ψηφίσουμε μαζί. Πρόκειται για τροπολογίε 797-42-55, 779-42-37, 780-42-38 και 773-42. Συμφωνείτε να τις ψηφίσουμε μαζί? Ωραία. Είναι κατά η συγκίτρια. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Καμία. Απορρίπτονται. 19.03.01.05. Τροπολίγιο 877 τώρα. Κατά η συγκίτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 21.03.01.04. Τροπολογία 80.16. Και 42.90. Κατά η εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται. Γραμμή 210701. Τροπολογία 540. Κατά. Είναι η συγκίτρια. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 230202 τροπολογία. 79-73 και τροπολογία 42-48. Είναι κατά η Γενική Συγκήτρια. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φτάνουμε στα σχόλια τώρα. Θα ψηφίσουμε μαζί. Τις γραμμές τις έχετε μπροστά σας. Τροπολογίες 43, 37, 36, 35, 34, 33, 32... 43, 31, 43, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 Μην τις διαβάζω όλες τις γραμμές έτσι. Υπέρ η συγκίτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δύο ψήφοι κατά. Εγκρίνονται λοιπόν. Συνεχίζουμε με τις παρατηρήσεις. Τώρα χωριστές ψηφοφορίες. 05, 01, 04, 03 γραμμή. Έχουμε την τροπολογία 41, 37. Είναι κατά η Γενική συγκίτρια. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13.05.60.01. Τροπολογία 170. Υπέρ, εισηγήτρια. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Ούτε κατά, ούτε αποχές. Εγκρίνεται. 19.02.02. Τροπολογία 374. Υπέρ η συγκεντρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο. Εγκρίνεται. Γραμμή 19.03.01.04. Τροπολογία 773. Υπέρ παρακαλώ. Η συγκέντρια είναι κατά. Έτσι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται. Γραμμή 19.03.01.05.877 877 τροπολογία. Η συγκέντρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19.03.01.06. Τροπολογία 176. Η συγκέντρια είναι κατά. Υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, αφού θέλετε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις σοφορίες. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ, 11 κατά και 2 αποχές. Περνάμε τώρα στη γραμμή 19.03.01.07, τροπολογία 157. αφού εγκρίναμε προηγουμένως μπορούμε να το ψηφίσουμε τροπολογία που είναι, οι οποίες είναι υπέρ ο 157 και 43-43 κατά κανείς αποχές 2, 3 εγκρίνονται 20.02.01 τροπολογία 3024 η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Καμία. Εγκρίνεται. Σχόλια που ψηφίζονται χωριστά τώρα. Γραμμή 220201, το απολογία 345. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 ψήφοι υπέρ, 16 κατά. Γραμμή 210204, τοπολογία 333. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Ε, είναι κατά, συγγνώμη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Καμία. Απορρίπτεται. Στην ίδια γραμμή. Τροπολογία 173. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21.02.07.01. 307 τροπολογία. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ κατά εγκρίνεται διορθώνει ο πρόεδρος απορρίπτεται 307 θέση γραμμή 210208 τροπολογία 648 και το τροπολογία 377 η εισηγήτρια είναι υπέρ ποιοι είναι υπέρ κατά τρεις ψήφοι κατά δεν υπάρχουν αποχές εγκρίνεται γραμμή 21-02-51-04-08-09 ε, η συγκίτρια είναι υπέρ θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 16 υπέρ 14 κατά 3 αποχές. 04, 40.48 η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, καμία. Απορρίπτεται. Γράμμη 21.03.02.03 απολογίες 180 και 634 η είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Στην ίδια γραμμή 175 η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές μία αποχή. Εγκρίνεται η τροπολογία. 21.04.01. 174 το υπολογία. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω κατά, δεν υπάρχει εποχή. Εγκρίνεται. Στην ίδια γραμμή. Οι είναι 614 και 379. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές 2 εγκρίνεται 21.08.02 γραμμή 323 τροπολογία εισηγήτρια είναι υπέρ ποιοι είναι υπέρ κατά 4 ψήφοι κατά εγκρίνεται Γραμμή 22.02.03.01 Τροπολογία 4062 Η εισηγήτρια είναι κατά Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δύο αποχές απορρίπτεται επτά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ισοψηφία 15-15. 22-03-01. Τροπολογία 4010. Η είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην ίδια γραμμή, τροπολογίες 172, 4186 και 728 με μια προφορική τροπολογία που προσθέτει and increase by 300.000 euros. Διορθώνει ο πρόεδρος, διαγράφει αυτή την φράση and increase by 300.000 euros. Ψηφίζουμε. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεν υπάρχουν. Εγκρίνεται. 23.09.06.01. Το υπολογείο 40.47. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ της τοπολογίας. Κανείς. Φαντάζομαι πολλοί θα ψηφίσετε κατά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελειώσαμε με την κατηγορία 4. Προχωρούμε στα πιλωτικά και προπαρασκευαστικές δράσεις. Συσυγήτρια. Έχετε κάτι να πείτε. Όχι. Ευχαριστώ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι όπως ξέρετε το να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα πίνακα με τα πιλωτικά και, τα, και τις προπαρασκευαστικές δράσεις προσπαθώντας να βρούμε ισορροπίες μεταξύ κατηγοριών, μεταξύ πιλωτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων και μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των επιτροπών είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει να κάνει κάποιος. Ελπίζω να καλύφθηκαν όλοι. Δεν μπόρεσα να βάλω πολύ περισσότερα πιλωτικά σχέδια και βασικές δράσεις από αυτές που είχαν προτείνει οι βουλευτές. Προφανώς όλα είναι ενδιαφέροντα. Δυστυχώς ωστόσο πρέπει να κρατήσουμε κάποια ανώτατα όρια για να καλύψουμε περισσότερο τον πίνακα. Ψηφίζουμε ε, συλλογικά όλα για το συμβαστικό κείμενο. Εισηγήτρια. Μια διευκρίνηση να κάνω μόνο. Λαμβάνοντας υπόψη το πώς ψηφίσαμε για τη μεταφορά κάποιων γραμμών στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης απελευθερώσαμε κάπου περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ ε, στην κατηγορία Α, 1α και μπορούμε να περάσουμε από την 3 στην 1α ένα πιλωτικό σχέδιο που ήταν Social Security Gap. Πιο λογικό ήταν να είναι στην 1α λόγω των περιορισμών ωστόσο ανωτά των ορίων την περάσαμε στην 3 όπου είχαμε περιθώριο. Με το κόψιμο τώρα μισού εκατομμυρίου μπορούμε να τα ξαναπεράσουμε, να ξαναπεράσουμε αυτό το πρόγραμμα στην 1α που είναι και πιο λογικό. Αλλάζεται λοιπόν το συμβιβαστικό κείμενο. Κύριε Ντεπρέ, δεν κατάλαβα μπορεί να επαναλάβει η Γενική συγγέντρη. τι είπε, γιατί είχα φερθεί. Ναι, λέω, ψηφίσαμε πριν λίγο να μεταφέρουμε από την κατηγορία 3 στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης ένα ποσό. Έχουμε 500.000 ευρώ στην κατηγορία 1α και έχουμε ένα πιλωτικό σχέδιο που μπορούμε να το περάσουμε εκεί. Αυτό λέω. Νομίζω ότι είναι σαφές για όλους μας. Ψηφίζουμε με άπαξ. Ποιοι είναι υπέρ της έγκρισης των θέσεων κατά εγκρίνεται Προχωρούμε λοιπόν στα άλλα τμήματα. Δίνω το λόγο στην κυρία Χολμάγερ, να θέλει να δώσει κάποιε διευκρινήσει. πριν ψηφίσουμε. Πολύ σύντομα. Δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με χθε. Τα στοιχεία είναι ίδια. Να εξηγήσω μόνο ότι μετά τον αφού ε, υιοθετήσαμε την θέση του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό, πρέπει να ψηφίσουμε τρεις τροπολογίες της EFDD. Στο, στο voting list φαίνεται ότι είναι τροπολογία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Δεν ισχύει αυτό. Είναι τροπολογία του EFDD. γιατί με ρωτήθηκα για ποιο λόγο απορρίπτουμε τροπολογίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Δεν είναι όμως ε, αλήθεια αυτό. Δεν κάναμε κάποια ψηφοφορία για το maintenance και το cleaning, αλλά ε, αναφερόμαστε ε, σε όσα συζητήσαμε στην Επιτροπή στους, με τους συντονιστές. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές. Merci, Madame le rapporteur. Donc, Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε. αποκατάσταση των πιστώσεων του σχεδίου προπολογισμού όπως έχει υποβληθεί από την Επιτροπή με κάποιες προσαρμογές στις οποίες επανέλθουμε. Υπέρ. Κατά. Έξι. Άρα περνάει. Τώρα υπάρχει μια προφορική τροπολογία της εισηγήτριας στη γραμμή 403 και στην γραμμή 101 η 403 είναι να δοθούν 3 εκατομμύρια και στην 101 να αφαιρεθούν 3 εκατομμύρια για να υπάρξει η ισορροπία μεταξύ του πλήν και του συν. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Θα γίνει ηλεκτρονικό έλεγχο καλύτερα. Άρχεται την ψηφοφορία. ψηφοφορία. ψηφοφορίας. 25-9. Διορθωτική επιστολή. της διεύθυνσης του Κοινοβουλίου. Έχετε τις λεπτομέρειες εδώ. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Έξι κατά. Διορθώνεται. Ε, εγκρίνεται η διορθωτική επιστολή. Τώρα προχωρούμε σε χωριστή ψηφοφορία. Γραμμή 1000. Τροπολογία 8019 και 4293. Όμοιες. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 1006. Τροπολογίες 80-20 και 42-94 με το ίδιο αντικείμενο. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στη γραμμή 1200, τροπολογία 8021 και 4295. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. απολύπτεται Γραμμή 1402. 80-22 και 42-96. Δεν τις θέλει η συγκεντρία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Στη γραμμή 2105. Το 83 83-92. Η συγκεντρία είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται στη γραμμή 400 τροπολογία 314 η κατά ποιοι είναι υπέρ τρεις ψήφοι κατά κατά αποχές δεν υπάρχουν. Γραμμή 400. 83-94. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι πέρα. Ποιοι είναι κατά. Έχει απορριφθεί. Τελειώσαμε. Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμβούλιο, τμήμα 2. Στην γραμμή 2010, λέει ο πρόεδρος. Ligne 2010, ligne 2200, ligne 2202. 2010, 2200, 2202. Τροπολογίες 2100, 2102 που είναι αντικείμενο 41-73 και 41-72 που ψηφίζονται ομού. Ποιοι είναι υπέρ. Η εισηγήτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ των τροπολογιών τώρα. Κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. Απορρίπτουν οι τροπολογίες. Προχωρούμε. Δικαστήριο. Τμήμα 4. Πρώτα, το συμβιβαστικό κείμενο Α. Δημιουργία 12 συμπληρωματικών θέσεων. Η εισηγήτρια είναι υπέρ, βεβαίως. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης, σηκώστε τα χέρια σας. Je vous remercie, contraire. Κατά. Αποχές. Τρεις. Εγκρίνεται. Άρα θα υπάρξει αύξηση του, σε καλύτερο, θα είναι επίπεδο ανταγωνισμό για, να για να βελτιώσει την ενιαία αγορά. Εννέα δικαστές τώρα για το δικαστήριο, η γενική η συγγήτρια είναι υπέρ. Κατά. Τη συμβαστική Β. Εγκρίθηκε. Σχόλια. Στην γραμμή 1406 η 2203 τροπολογία η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Ψήφι κατά. Όχι, μία αποχή, δύο αποχές. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. Τμήμα 6. Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή. ΕΟΚΕ. Συμφωνία Συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ υπάρχει ένα συμβιβαστικό κείμενο και μία ψηφοφορία ομού. Η συγκεκριμένη είναι υπέρ. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δέκα. Εγκρίνεται. Προχωρούμε. προτάσεις της εισηγήτριας για το τμήμα 7. Υπάρχει μια ψηφοφορία για το συμβαστικό κείμενο όπου υπάρχει υποστήριξη της εισηγήτριας. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίνεται το πακέτο. χωριστές ψηφοφορίες. Στη 1004 καταρχάς η τροπολογία 7600. Η συγκίτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για αυτή την τροπολογία, άρχιτη ψηφοφορία. Scrutin est clos. Le vote est actif à 22 voix contre 12. Ε, 22-12. Στη γραμμή 2-64 υπάρχει τροπολογία 25-03 όπου η συγγητής η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 23-12 εγκρίνεται στη γραμμή S7-S1 μια πρώτη τροπολογία 4036 και μια άλλη που έχει τον ίδιο αριθμό Πάντω και με τις δύο η συγκίτρια είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Τι, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τμήμα 10. Εξωτερική, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Τρεις τροπολογίες έχουμε. Στις θέσεις 3001, 3003 και 3004. Η 2809 τροπολογία. Η 2810 και η 2811. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε ομού. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά αποχές καμία εκκρίνονται. Eh bien, Τελειώσαμε με αυτό το τμήμα, δηλαδή τα άλλα τμήματα του προπολογισμού. Τώρα έχουμε τις πληρωμές. Για τις πληρωμές έχουμε πρώτα απ' όλα ψηφοφορίες ομαδοποιημένες, μπλοκ. Πρώτη ομάδα που θέλει να επανέλθουμε στα ποσά του πρώτου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εισηγήτρια είναι Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Πέντε. Λοιπόν. Αποχές δεν έχουμε. Α, κύριε Ντεπρέ, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, πρόεδρε, πριν ψηφίσουμε το, τη δεύτερη ομάδα και την τρίτη ομάδα, θα είδατε ότι για την πρώτη ομάδα δεν βάζουμε κανένα πρόβλημα. Συμφωνούμε. Εξάλλου για μας μόνο το επίπεδο υποχρεώσεων ήταν ε, που δεν το θέλαμε έτσι ακριβώς όπως αυτό που εγκρίθηκε, αλλά ψηφίζουμε υπέρ για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, γιατί πρέπει να φανούμε ενωμένοι απέναντι στο Συμβούλιο. Για το 3 θέλω να υπενθυμίσω ότι είχαμε υποβάλει ενστάσεις όσον αφορά την χρησιμότητα σε αυτό το στάδιο να ξοδέψουμε ολόκληρο το contingency και ζήτησα από την ομάδα μου ναι, να το υπερψηφίσει, αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ, δεδομένης της ευαισθησίας που έχει η ομάδα μου, ότι θα ακολουθήσει γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι η καλύτερη περίπτωση. Πάντως εγώ θα στηρίξω την απόφαση της Επιτροπής μας, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να φανούμε ενωμένοι, αλλά δεν μπορώ να σας εγγυθώ για το τι θα ψηφίσει η ομάδα μου. Πρόεδρος, ωραία, όλοι λίγο πολύ νιώσαμε περίεργα για να ψηφίσουμε εδώ, γιατί το βασικό πρόβλημά μας είναι αυτά τα ποσά που έπρεπε να έχουν πληρωθεί και δεν έχουν πληρωθεί. Ελπίζουμε και θα επιμείνουμε στο Συμβούλιο και την Επιτροπή τις επόμενες μέρες για να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν εξαρτάται το θα ψηφίσουμε εμείς εδώ απαραίτητα, οπότε με τη δικιά σας την στήριξη πρέπει να δώσουμε αυτό τον αγώνα. Λοιπόν, ψηφίσαμε για το 1. Ομάδα 2 τώρα. Υπέρ η συγγήτρια. Ψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Κατά. Πέντε ψηφίκατα κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία αυτή, το μπλοκ 2 δηλαδή. Και τώρα η τρίτη ομάδα, μπλοκ 3, που θέλει να έρθουμε σε επίπεδο πολύ παραπάνω από τα αρχικά ποσά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπέρ η Γενική Συγκήτρια. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Πέντε. Συνεπώς, ψηφίσαμε τις τρεις αυτές ομάδες, είναι η διαπραγματευτική μας θέση, έτσι. Ερχόμαστε τώρα στις χωριστές ψηφοφορίες, 040260, ...2014-2020 υπέρ κατά αποχές Δεν έχουμε αποχές. Απορρίπτεται. Γραμμή 040261. 2014-2020 κατά η Γενική Συγγήτρια. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν έχουμε. Απορρίπτεται. Γραμμή 040262. 2014-2020. Κατά η Γενική Συγκήτρια. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τελειώσαμε. Μέχρι αύριο το βράδυ κανονικά θα ήμασταν εδώ. Η κυρία Κοζαμπάλα, οι συντονιστές, η κυρία Χολμάγερ ετοίμασαν τόσο καλά την ψηφοφορία. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω, όπως επίσης και τη γραμματεία μας και την Μάνικα Στράσερ, την επικεφαλής της γραμματείας, για την εξαιρετική δουλειά τους αυτή την ψηφοφορία. Το λέω έτσι αυθόρμητα αυθορμητισμό που χαρακτηρίζει τους νέους εδώ στην Επιτροπή. Παρακαλώ την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Για να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να καθίσουμε και να σκεφτούμε καλύτερα το τι ψηφίσαμε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην Επιτροπή μας, γιατί νομίζω ότι κάναμε, κάνουμε έτσι μια πρόταση διαπραγμάτευσης ανοιχτή. Διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, όμως πέρα από αυτά τα οποία ψηφίσαμε, γιατί τώρα θα μπούμε στις διαπραγματεύσεις και τώρα είναι που θα καταλήξουμε στα τελικά ποσά. Νομίζω ότι πετύχαμε αυτό που θέλαμε μέχρι τώρα και εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συντονιστές και όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες. Ξέρουμε πόσο περίπλοκη είναι όλη αυτή η διαδικασία. αλλά οι συντονιστές βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να επιτευχθούν οι συμφωνίες και όπως είπατε και εσείς ιδιαίτερα ευχαριστούμε τη γραμματεία. Είναι τόσο δύσκολο να δουλέψει κανείς με όλες αυτές τις τροπολογίες κάθε τέταρτο να αλλάζει κάτι γιατί αλλάζουν οι συμφωνίες μεταξύ μας και ο κατάλογος ψηφοφοριών, οπότε μπράβο στη γραμματεία που μας διευκόλυνε τόσο πολύ τη δουλειά. Συγχαρητήρια και μια που είναι εδώ, η Μόνικα και ο Χόλγαν, αλλά και όλους τους υπόλοιπους έτσι, που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω ότι μετά από τη δουλειά αυτή το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτός είναι και ο πότερος στόχος μας. Ε, Πρόεδρος, όντως, γιγάντιο έργο. Γι' αυτό και ιδιαίτερε ευχαριστίες μου και προς τη Γενική Συγκίτρια και προς τους ηγητές των άλλων τμήματων, προς τους συντονιστές, όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής. Στη Γραμματεία επίσης, για το αξέρετο έργο της. Πραγματικά νιώθω ευγνωμοσύνη και θαυμασμό. Καρπός τώρα των ψηφοφοριών αυτών είναι να βάλουμε τον πύχη σε ένα καλό επίπεδο διαπραγματεύσεων. Ψηλό. Να δούμε τώρα το Συμβούλιο από τη δικιά του την πλευρά και η Επιτροπή τι θα κάνουν. Γιατί θέλουμε να λύξει αυτό το πρόβλημα με τις πληρωμές που έχουμε, που είναι αφόρητο και που δίνει μια πέσια εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί χρωστάμε χρήματα στις περιφέρειες, στις τοπικές δικήσεις που δεν παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Είναι και θέμα ανθρωπιστικών οργανώσεων που δεν πληρώνονται, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων. Εμείς που θέλουμε να δώσουμε όθεση στην ανάπτυξη, καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια καθυστέρηση είναι απαράδεκτη. Ψάχνουμε λύσεις λοιπόν. Τώρα θα δούμε Οι ψηφοφορίες στις οποίες καταλήξαμε, το αποτέλεσμά τους ε, βασικά, δείχνει πόσο μεγάλη, υπάρχει, μεγάλη ανάγκη υπάρχει να βρεθούν λύσεις και να έχουμε κάποια περιθώρια. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να φαντάζεστε ότι τα 300 δισεκατομμύρια που υποσχέθηκαν θα έρθουν το 2016, το 2017 και μετά. Όχι, τώρα. Και τώρα πρέπει να σβήσει η φωτιά που έχει ανάψει. Βρισκόμαστε σε έκτακτη ανάγκη. Ψηφίζοντας δείξαμε ότι οι προσδοκίες μας είναι πάρα πολύ ψηλές. Τώρα περιμένουμε να δούμε σε τι συμβασμό θα καταλήξουμε με το Συμβούλιο. Στόχος είναι η σύγκληση βέβαια. Πρέπει να βρούμε τώρα πώς θα το πετύχουμε αυτό. Και ξέρουμε όλοι ότι ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Κατόπιν όλων αυτών, α επωφεληθούμε από τον ελεύθερο χρόνο που μα μένει, μια που είχαμε προβλέψει να συνεδριάσουμε σήμερα το απόγευμα και αύριο ενδεχομένω. Οπότε μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε τι ακρόασει των ε, μελλοντικών επιτρόπων και να ετοιμάσουμε και τη δικιά μα ακρόαση με την κυρία Γεώργιεβα που προβλέπεται για την 5η το μεσημέρι 2 Οκτωβρίου στη 1.30. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε μήπως κάτι άλλο, ερωτήσεις, κάτι, όχι, ωραία. Κυρίσω τη λήξη της συνεδρίασης.